Αρχίζουμε με τις επεξηγήσεις ψήφου στην έκθεση Μπροκ και Γκολτιέρη. Πρώτη η κυρία Οβίρ για ένα λεπτό. Juhataja, Euroopa ühises tegutsemises on väärtus. Euroopa saab põhimõtteliselt või Eurotsoon saab põhimõtteliselt... Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε Ξέρετε πως ε, η Ευρωζώνη μπορεί να πάει προς δύο μόνο ή να ενισχυθεί ή να καταρρεύσει. Στην ε, τωρινή οικονομική κατάσταση πρέπει να αντιδράσουμε γρήγορα. Εγώ υποστηρίζω το μηχανισμό σταθερότητας και την ε, έκθεση αυτή γιατί δημιουργεί ένα νομικό πλαίσιο για την εφαρμογή του μηχανισμού αυτού. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χτες ε, ψηφίσαμε για το μόνισμο μηχανισμό σταθερότητας ε, και δεν τα καταφέραμε. Η τροπολογία 33 αποσύρθηκε που θα μας έδινε δυνατότητα αγορών στις δευτερογενείς αγορές και ε, δεν μπορέσαμε να λάβουμε τις σκληρές αποφάσεις. Είναι σκληρές αποφάσεις αλλά θα έκριναν το μέλλον ή την αποτυχία της Ευρωζώνης χώνουμε το κεφάλι μας στην άμμο σαν τους τρουθοκάμιλους. Έχουμε εκτός από νομισματική κρίση και τραπεζική κρίση και κρίση δημοσίου χρέους. Και εξακολουθούμε στις πληγές να βάζουμε χαζαπλάστ. Η ίδια μου η χώρα, η Ιρλανδία, έχει αβάσταχτο βάρος γιατί Αγγλία, Γαλλία και γερμανικές ε, τράπεζες δεν είχαν επιτήρηση και λειτουργούσαν ω καζίνο. Πλέον δεν μιλάμε για δημόσιο χρέο, μιλάμε για χρέο των πολιτών και όλα αυτά έγιναν κάτω από τη μύτη τη Ευρωπαϊκή Κρατική Τράπεζα με τελείω απαράδεκτα επιτόκια. Και όλα αυτά θα τα πληρώσουν οι Ιρλανδοί πολίτε. Κανεί δεν αντιμετωπίζει την πραγματικότητα. Δεν είναι βιώσιμο το χρέος. Χρειάζεται μεγάλη αναδιάρθρωση. Ευχαριστώ. Χρειαζόμαστε ένα μόνιμο μηχανισμό διαχείρισης των κρίσεων στην Ευρώπη για να παρεμποδίσουμε τουλάχιστον να αντιμετωπίσουμε μελλοντικέ οικονομικές κρίσεις. Τα πράγματα θα χειροτερέψουν αν δεν είμαστε προσεκτικοί και είναι θλιβερό το ότι αυτός ο μηχανισμός προγραμματίζεται εντελώς εκτός των οργάνων της Ένωσης. Θα πρέπει να παίρνουμε μέρος στον προγραμματισμό όσο πιο πολύ γίνεται κι εμείς. Βέβαια είναι καλό το ότι χώρε όπως η Σουηδία και η Βρετανία βρίσκονται εκτός της Ευρωζώνης αν θα μπορούσαν και αυτές να πάρουν μέρος. Χρειαζόμαστε πιο επαρκή συντονισμό των οικονομικών πολιτικών μα στην Ευρώπη και όταν υπάρχουν κυρώσεις να αποφασίζονται από την Κομισιόν και να είναι αυτόματος και χωρίς συζήτηση και παζάρια. Ευχαριστώ. Thank you, Mr. President. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μετά από 12 χρόνια ευρωβουλευτής τίποτα δεν θα με ξάφνιαζε νόμιζα, αλλά σοκαρίστηκα από τον τρόπο με τον οποίο ο κύριος Μπρόκ εισήγαγε την έκθεση του χθε. Με σοκάρισε και η έπαρση και ότι είναι άσχετο με την πραγματικότητα και ο, περιορισμό, και ο περιφρόνης κοινής νόμης. Αλλά είπε ότι πρέπει να αποφύγουμε την διαδικασία ενεθόρησης συνθήκης γιατί διαφορετικά αυτό μπορεί να οδηγήσει σε δημοψήφισμα σε μερικά κράτη-μέλη. Βλέπετε την περιφρόνηση εκ μέρους των Ελλήνων της Ένωσης απέναντι στους πολίτες, την κοινή γνώμη, τη μεταχειριζόμαστε όχι έναν τρόπο για να αλλάξουμε κατεύθυνση, αλλά σε ένα εμπόδιο που πρέπει να υπερπηδηθεί. Θυμίζω, θυμάμαι του συμπατριώτες του κυρίου Μπροκ όταν είχαμε τα γεγονότα στο Ανατολικό Γεγολίνο. Κάποιος είπε εύκολο ήταν να, πιο εύκολο θα ήταν να διαλύσουμε το λαό. Ο κύριος Καμάλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ένα από τα εγγενή προβλήματα ενός ενιαίου νομίσματος με πολλά κράτη-μέλη και διαφορετικούς οικονομικούς κύκλους είναι πως καλό είναι να έχουμε ένα επιτόκιο εάν ε, έχουμε διαφορετικά έξοδα. Και βλέπουμε το αποτέλεσμα τώρα, βλέπουμε τα προβλήματα της Ευρωζώνης. Αλλά πέρα από αυτό, οι κυβερνήσεις πρέπει να αντιληφθούν πως δεν μπορούν να ξοδεύουν περισσότερα από τα έσοδά τους. Και όταν το κάνουν αυτό και μαγειρεύουν τα βιβλία και δεν εκπληρώνουν τον ρόλο τους ως ε, οικονομική διακυβέρνηση, μπλέκουν και οι άλλοι. Και πρέπει να είμαστε σαφεί πω εάν είναι κάποιο στην Ευρωζώνη, βεβαίω θα είναι ισχυρή Ευρωζώνη, ειδικά για τα μέλη εκτό Ευρωζώνη. Θέλουμε να συνεχίσουμε να εμπορευόμαστε με τι χώρε τη Ευρωζώνη και δεν εποφελούμαστε από το ασθενέ ευρώ. Αλλά οι ίδιες οι χώρες ε, εκείνες πρέπει να λύσουν τα προβλήματά του και να μην βασίζονται σε άλλου. Σα εύχομαι καλή τύχη και σα παρακαλώ μην ξοδεύετε περισσότερα από όσα έχετε. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ξεκαθαρίσω εξ ονόματος των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών πως είμαστε υπέρ του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας ε, που συστήθηκε. Αλλά καταψηφίσαμε την έκθεση Μπροκ Γκουαλτιέρη γιατί αυτή η γνωμοδότηση δεν συμφωνούσε με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου. Αυτό το οποίο ήθελε η έκθεση αυτή ήταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Κομισιόν να εμπλακούν ουσιαστικά σε έναν διακυβερνητικό μηχανισμό. Και θα πρέπει να είναι διακυβερνητικός αυτός ο μηχανισμός λόγω των τεραστίων ποσών που έχουν δεσμευτεί και οι εθνικοί υπουργοί που λογοδοτούν στα εθνικά κοινοβούλια είναι οι σωστοί γραμμή ευθύνη. Βεβαίω, πίσω από όλη αυτή την κρίση δεν είναι το πρόβλημα με το ευρώ, αλλά πρόβλημα με τι κυβερνήσει που ξοδεύουν πάρα πολλά λεφτά των φορολογουμένων. Ευχαριστώ. Περνάμε τώρα στην έκθεση Ζασάντα, ο κύριος Καμάλ για ένα λεπτό. Mr. Kamal, go ahead. Thank you very much. Um, I welcome... Ευχαριστώ επικροτώ τη δεύτερη φάση, τα πορίσματα της δεύτερης φάσης της ε, συμφωνίας αυτής. Είναι μια πολύ καλή λύση, αλλά όσοι από εμά θέλαμε περισσότερη φιλελευθερωποίηση και να φύγουμε από τον προστατευτισμό που ακόμα μπλοκάρει αυτό τον κλάδο από πολλές. Θα ήθελα οι Ηνωμένες Πολιτείες να άρουν τα εμπόδια και τους περιορισμούς σε ξένη ιδιοκτησία και ε, ε, μετακινούμενοι να επωφεληθούν από τους ανοιχτούς ουρανούς. Συγχαίρω την Τζάκη Φώστερ που είναι εμπειρογνώμων στο θέμα αυτό. Έχει δουλέψει και για τις μεταφορές και είναι ενεργό μέλος στην Επιτροπή Μεταφορών. Αλλά μόνο αν συνεχίσουμε να πιέζουμε περαιτέρω φιλελευθερωποίηση και στις ΗΠΑ και στι αναδυόμενε αγορές της Ασία και επικροτώ την κίνηση σήμερα σχετικά με τη συμφωνία με το Βιετνάμ αν συνεχίσουμε έτσι να έχουμε πρόσβαση στις αναπτυσσόμενες αγορές του κόσμου. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σαρλάκη, για ένα λεπτό. Not in the room. Έκθεση Μπαλζάνη. Ο κύριος Ντεάντζελης, ένα λεπτό. Mr. De Angelis, one minute. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν ευχαριστώ την εισηγήτρια Μπαλσάνη για την άριστη εργασία της. Τέσσερα είναι τα σημεία της έκθεσης πρωτοβουλίας που θεωρώ σημαντικά. Το πρώτο, γενικά, σαφής έκκληση στον προπολογισμό της Ένωσης και την αναδιαναμερική του φύση ως βάση της Ευρωπαϊκής Αλληλεγγύης. Δεύτερο, το ειδικό πρόγραμμα με βάση την αρχή όπου ειδικά στον τομέα της συνοχής θα πρέπει να επιληθούν όχι με τον τρόπο που προτείνει το Συμβούλιο. Τρίτο, αμφιβολίες σχετικά με το αποτελεσμό του κριτήριου προβλεψιμότητας με βάση την προηγούμενη οικονομική άσκηση και καλείται η Κομισιό να κάνει προτάσεις για τη δημιουργία νέων πόρων. Το τέταρτο, οι νέοι πόροι θα πρέπει να έχουν στόχο να καταπολεμηθεί η κρίση με συγκεκριμένη δέσμευση υπέρ πολιτικών καινοτομία, έρευνας και οικονομικής παραγωγικής ανάπτυξης και για την απασχόληση στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ιακολίνο. Πρόεδρε, σε μια τόσο σημαντική φάση ένα τέτοιο έγγραφο θα πρέπει να κριθεί με βάση τα κριτήρια της κοινής λογικής. Την υποστήριξουμε την, την στρατηγική του 2020 είναι μια έκφραση και αξιοπιστίας και συνοχής εκ μέρους του Ευρωκοινοβουλίου. Μερικά κριτήρια και κατευθυντήριες γραμμές θα έπρεπε περαιτέρω να ενισχυθούν μέσω ενός καταλόγου προτεραιοτήτων για παρεμβάσεις σήμερα σε μια τόσο δύσκολη στιγμή όπου κυρίως στη Μεσόγειο αλλά και στην Ιαπωνία οι δυσκολίες συνδέονται με μια πραγματικότητα η οποία αλλάζει πολύ γρήγορα υπάρχει ανάγκη το Ευρωκοινοβούλιο να είναι φερέγγιο με κύρος να δίνει απαντήσεις υπέρ της οικονομικής ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας, της βιωσιμότητας με έξυπνο τρόπο. Ευχαριστώ. Μποργέζιο, ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σε μια τόσο λεπτή φάση όπως είπε ο συνάδελφος πριν όσα αφορά τα οικονομικά των κρατών μελών κρούω τον κόδυνα του κινδύνου για κάτι που συζητιέται στην Επιτροπή Προπολογισμών. Μια περίπτωση θα την έλεγα αν εγκριθεί το τεράστιο κόστος που προβλέπεται για το σπίτι της ευρωπαϊκής ιστορίας το κτίριο Eastman είναι η διοκτησία μας, αλλά μόνο για τις διαπάνες αναδιάρθρωσης του κτιρίου προβλέπονται 26 και 31 εκατομμύρια ευρώ. 3,3 μόνο πάνε για τα σχέδια. Πάνω από 3% λειτουργικά. Για το προσωπικό 50 άτομα, 3,2 εκατομμύρια ευρώ. 2 εκατομμύρια για την ασφάλεια μόνο για τη διαχείριση 13,45 εκατομμύρια ευρώ. Πρέπει να δώσουμε το παράδειγμα σχετικά με τις πολυτελείς δαπάνες. Θα ήταν έσχος κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να υποβάλω τρεις παρατηρήσεις για, για το προσχέδιο προϋπολογισμού του 2012. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό που σε τόσο πρόωρη φάση ασχολούμαστε με αυτό για να αποφύγουμε τη θλιβερή εικόνα που δώσαμε τα τρία θεσμικά όργανα στον προϋπολογισμό του 2011. Και είμαι ιδιαίτερη περήφανος που δεν προβλέπονται συμπληρωματικά κονδύλια για τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Ελπίζω να συνεχιστεί αυτό. Η κυρία Οβίρ για ένα λεπτό. president! Ευχαριστώ. Η νόμιμη μετανάστευση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας και προωθεί την ανταγωνιστικότητά μας. Ένα από τα προβλήματα όμως οφείλεται στο, νομικό καθεστώς που ισχύει για τους μετανάστες μάλλον το γεγονός ότι δεν έχουν τέτοιο νομικό καθεστώς και υφίστανται διακριτική μεταχείριση. Είναι κρίμα που στον 21ο αιώνα μερικοί άνθρωποι δουλεύουν εδώ σε συνθήκες υλωτίας. Όλοι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να τη χάνουν ίσης μεταχείρισης σε μια νέα ευρωπαϊκή αγορά. Η έκθεση αυτή συμπληρώνει την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Γι' αυτό και είμαι υπέρ τη δημιουργία ενό νομικού πλαισίου που θα γεφυρώνει το κενό που υπάρχει μέχρι στιγμή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η διοικητική απλούστευση και η της πρόσβασης σε σχετικές πληροφορίες είναι εργαλεία κατάλληλα έτσι ώστε η αγορά εργασίας στην Ευρώπη να γίνει πιο ελκυστική για τους εργαζόμενους τρίτων χωρών. Η σύστηση μιας ενιαίας διαδικασίας ετήσεω και ένας τίτλος που ανακαλύπτει και την άδεια παραμονής και την άδεια εργασίας με μία διοικητική πράξη θα απλοποιήσει και θα εναρμονίσει τις διατάξεις που ισχύουν τώρα από χώρα σε χώρα. Έτσι θα είναι πιο σαφής η διαδικασία και για τον μετανάστη και για τον εργοδότη. Και ταυτόχρονα θα διευκολυθούν οι έλεγχοι για την νομιμότητα παραμονής και απασχόλησης. Η ενιαία διαδικασία θα επιτρέψει να μειωθούν οι ανισότητες των δικαιωμάτων μεταξύ των πολιτών της Ένωσης και των πολιτών τρίτων χωρών. Γι' αυτό ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος συναδέλφου Ματιού. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ψήφισα κατά της πρότασης οδηγίας αυτής γιατί πρέπει να εφαρμόσουμε μία ενιαία προσέγγιση στην ενιαία άδεια Θα πρέπει να δημιουργηθούν δηλαδή κανόνες ε, για τους υπηκός τρίτων χωρών που βρίσκονται στις, ε, σε ένα κράτος μέλος. Ε, η νομική βεβαιότητα και η διαφάνεια κατά την λήψη των αποφάσεων και την επεξεργασία των αιτήσεων είναι επίση αναγκαία γιατί θα πρέπει να εξετάζονται αντικειμενικά. Η ίδια μεταχείριση πρέπει να υπάρχει σε όλους τους τομείς της κοινωνίας και να υπάρχει σωστή ε, νομοθεσία. Επειδή λοιπόν αυτά δεν υπήρχαν ε, στην ε, οδηγία δεν το θεωρώ στο αυτό το οποίο ήθελαν τα δεξιά κόμματα. Ο κύριος Στάκουλα, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Εδώ μιλούμε για τα δικαιώματα των αλλοδαπών εργαζομένων, των νόμων μεταναστών στην Ευρώπη. Θα πρέπει να αξιοποιηθούμε τα δικαιώματα των εργαζομένων υπηκών των χωρών μελών. Είναι ένα καλό σημείο αφετηρία η έκθεση αυτή. Θα πρέπει να καταβάλλεται ίσως μισθός για ίση εργασία και με τις ίδιες εργασιακές συνθήκες. Είναι πολύ καλή λοιπόν η έκθεση αυτή ω σημείο φετηρία, αλλά παρόλα αυτά δημιουργεί κάποιε ανησυχίε. Στο άρθρο 3 συγκεκριμένα, και σε κάποια εδάφια του άρθρου 3, θα πρέπει να μην ξεχνούμε και τους εποχιακούς ή προσωρινά εργαζόμενους, γιατί δεν θα πρέπει να τους ξεχνάμε. Θα πρέπει όλοι αυτοί οι άνθρωποι να έχουν πρόσβαση στα ίδια, στα ίδια δικαιώματα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ με τους ε, συναδέλφους εκείνους ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που λένε πως πρέπει να υπάρχει ίση μεταχείριση για εργαζομένους τρίτων χωρών που απασχολείται για παραπάνω από ένα έτος. Επίσης συμφωνώ με το ότι οι εργαζόμενοι που παραμένουν λιγότερο από έξι μήνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εργάζονται ε, πρέπει να έχουν μεταχείριση ίση όσον αφορά τις κοινωνικές παροχές. Ε, δεν ξέρω όμως ε, τι θα πρέπει να γίνει με την, απασχόλη, με την ασφάλιση ε, ασθένειας και ατυχημάτων. Και θα πρέπει να ισχύουν οι κανόνες του κράτους μέλους ε, αρκεί βεβαίως να το επιθυμεί και το τρίτο και η τρίτη χώρα. Ο κύριος Φόξ έχει ζητήσει το λόγο για την προηγούμενη έκθεση της κυρίας Μπαλτζάνη, την κατάρτιση του προπολογισμού του 2012. Έχετε το λόγο κύριε Φόξ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλωσορίζω το ότι ξεκινάμε προετοιμασίες τόσο νωρίς για τον προπολογισμό του 2012. Έτσι θα εξετάσουμε σωστά τα θέματα. Ένα από τα ζητήματα τα οποία συζητάμε συχνά εδώ πέρα σε αυτό το μικυκλίο είναι το θέμα της αλληλεγγύης. Ε, δείχνουμε αλληλεγγύη σε διάφορες ομάδες. Εγώ θα ζητήσω από το Κοινοβούλιο αυτό να δείξει αλληλεγγύη με τους φορολογουμένους, τους ε, ψηφοφόρους μας, γιατί δεν το έχουμε κάνει. Και στην εποχή λιτότητας πρέπει να επιδείξουμε αυτοσυγκράτηση, να δώσουμε το καλό παράδειγμα, παγώνοντας τους μισθούς και τα επιδόματα των Ευρωβουλευτών και των υπαλλήλων για το 2012, και να εγκαταλείψουμε σχέδια για το σπίτι της ευρωπαϊκής ιστορίας που θα κοστίσει εκατομμύρια ευρώ και για το οποίο δεν υπάρχει μακροπρόθεσμο σχέδιο χρηματοδότησης και πάλι οι φορολογούμενοι θα το πληρώσουν. Ευχαριστώ. Ο κύριος ένα Go ahead, Mr. Σε ποιο ψήφισμα να μιλήσω. Σουάμπ. Ευχαριστώ. Ο κατακαιρματισμός των νομοθετημάτων σε θέματα δικαιωμάτων των καταναλωτών αποτελεί, αποτελεί μεγάλο εμπόδιο και για την κτήση και για την πώληση διασυνοριακά και η δημιουργία μιας πραγματικής εσωτερικής αγοράς ε, ε, εμποδίζεται. Η πρόταση οδηγίας σήμερα που ξεκίνησε θα συμβάλλει στο να υπάρξει ένα σαφέ νομικό πλαίσιο στον αφορά τα δικαιώματα των καταναλωτών. Ευχαριστώ. Ο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Η έκθεση αυτή με βάση την αναθεώρηση των τεσσάρων οδηγιών που ισχύουν προτείνει να σταματήσει να ισχύει ένα πλαίσιο το οποίο δημιούργησε ένα σωρό εμπόδια μέχρι σήμερα στην εσωτερική αγρά. Ο στόχος είναι να βελτιωθεί η λειτουργία της για τον καταναλωτή και τις επιχειρήσεις αυξάντη την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και μειώνοντας την δισταγμό των επιχειρήσεων να λειτουργήσουν διασυνοριακά. Η πρόταση είναι πολύπλοκη, έχει πολλές λεπτομέρειες. Όλα αυτά συζητήθηκαν και από την προηγούμενη Γαλλική Προεδρία. Με την Επιτροπή Μπαρός όμως και την Επιτροπή Ρέντινγκ η πλήρης εναρμόνιση δεν θεωρήθηκε δόγμα και σωστά ξεκίνησε μια κίνηση με πιο συγκεκριμένη εναρμόνιση. Είμαι μεν ικανοποιημένο από το αποτέλεσμα, που το θεωρώ όμω μέτριο, είναι καρπός ενός συμβασμού προς τα κάτω και γι' αυτό εύχομαι η πρόταση αυτή να αποτελέσει αφετηρία για περαιτέρω εξελίξεις και γι' αυτό υποστήριξα αυτό το ψήφισμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο Λαβία για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ συνάδελφοι, ε, το κείμενο που ψηφίσαμε σύντομα βγήκε από μια πολύπλοκη διαδικασία που ξεκίνησε από το 2008 από μέρη στο κέντρο των καταναλωτή όσον αφορά τι πωλήσει ενεργειακές. Ο στόχος είναι να συμβάλλουμε σε μια καλύτερη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, περισσότερη κατανάλωση εκ μέρους του καταναλωτή και υποστηρίξη των επιχειρήσεων μας. Η οδηγία που ψηφίστηκε είναι η σύνθεση τεσσάρων ιδιών σχετικών που ίσχυαν μέχρι σήμερα και εκφράζει τη βούληση εναρμόνισης, την πειθαρχία που ισχύει σήμερα, αποφεύγοντας τον νομικό κατακαιρματισμό που δυστυχώς συχνά αποτελεί εμπόδιο και για τις επιχειρήσεις που στόχος τους είναι, είναι ανταγωνιστικές στη στην αγορά και για τον καταναλωτή. Γι' αυτό ψήφισα το ψήφισμα, υπερψήφιση του ψήφισμα αυτό. Ευχαριστώ. Κόμι, Ο κύριος Ρέπο, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η αναθεώρηση αυτής της οδηγίας ήταν μια χρονοβόρα διαδικασία και ο κίνδυνος ήταν να μην επιφέρουμε αλλαγές που θα υποβαθμίσουν το επίπεδο προστασίας στις σκανδιναβικές χώρες δημιουργών, επιβάλλοντας ένα συντονισμό προς τον ελάχιστο κοινό παρανομαστή. Οι συμφωνίες με τις οργανώσεις καταναλωτών θα πρέπει να προσανατολίζονται στις καλύτερες δυνατές ρυθμίσεις για αυτούς. Ας μην ξεχνάμε ότι η αγορά θα πρέπει να εξυπηρετεί τους καταναλωτές και όχι το αντίστροφο. Οπότε θα πρέπει να θεσπίσουμε σαφείς, απλούς και εύληπτους κανόνες για να προστατεύσουμε τα δικαιώματα των καταναλωτών. Νομίζω ότι είναι σωστή η απόφαση του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Η εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αναπτυχθεί εντυπωσιακά. Γι' αυτό καλό θα είναι να εξετάσουμε κατά πόσο πραγματικά εξυπηρετεί τα συμφέροντα και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των καταναλωτών. Η πρόταση αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών προκάλεσε ανάμεικτα συναισθήματα στις φιλανδικές οργανώσεις καταναλωτών έγιναν κάποιες διαμαρτυρίες και συγκεντρώθηκαν υπογραφές για το θέμα αυτό και μάλιστα επιβλήσαν και αναφορέ γιατί θεωρούμε ότι η πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αποδυναμώσει την προστασία των καταναλωτών στη Φιλανδία. Καταλήξαμε σε πολλέ συμβαστικέ λύσει που ήταν το αποτέλεσμα σφοδρή συζήτηση, αλλά ο συμβασμό δεν ήταν εύκολο. Δεν είναι αρκετά φιλόδοξη η τελική πρόταση. Και το βασικό πρόβλημα έγκυται στο ότι είναι πολύ δύσκολο να γίνει αντιληπτή από τις ε, οργανώσεις των καταναλωτών. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι να καταλαβαίνουν οι καταναλωτέ αυτή την οδηγία, αφού για αυτού έγινε. Ε, ευχαριστώ. Ε, Βεβαίω μίλησαν ήδη άλλοι δύο Φιλανδοί συνάδελφοι και η κυρία Γιατερμάκη εξέφρασε ξεκάθαρα τι απόψει μα για την οδηγία αυτή ανησυχούμε για το ότι υπάρχει κίνδυνος να εξασθενήσει η προστασία των καταναλωτών στη Φιλανδία και στις άλλες σκανδιναβικές χώρες. Υπάρχει επίσης ανησυχία ότι πολλές από τις διαδικασίες θα επιβραδυνθούν. Υπήρχαν πολύ προβληματικοί τομεί όταν το συζητούσαμε αυτό στην Επιτροπή και ελπίζω στην Επιτροπή όπου το αναπέμψαμε τώρα να μπορέσουμε να λύσουμε κάποια από τα δύσκολα αυτά θέματα. Παραδείγματο χάρη έχουμε τουριστικές επιχειρήσεις που τις βλέπουν έτσι πάρα πολύ αρνητικά στη Βόρεια Φιλανδία και δυσκολεύεται ο κόσμος ε, να κλείσει το μάτι ξενοδοχείου ή να κάνει τις κρατήσεις του γενικώς. Οπότε θα πρέπει να υπάρχει η προστασία αυτή κατά τρόπον ώστε να μπορεί ο κόσμος να ξέρει πώς θα χρησιμοποιήσει υπηρεσίες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θεωρώ πως η πρόταση αυτή η εναρμόνιση των ε, θεμάτων αυτών που κατακαιρματίζουν το ευρωπαϊκό εμπόριο είναι καλό. Θα πρέπει να υπάρχει ένα ευρωπαϊκό περιδικαίου αίσθημα του καταναλωτή, δηλαδή να είναι σίγουρος όταν αγοράζει κάτι μέσω διαδικτύου. Αυτό δεν είναι μόνο για την ασφάλεια του καταναλωτή, αλλά και για του παραγωγού. Χαίρομαι ιδιαίτερα για τις βελτιώσεις στις υποχρεώσεις ε, πληροφόρησης για τις ε, πωλήσει ε, πόρτα-πόρτα και για τις συμβάσεις εξ αποστάσεως. Θα πρέπει να δώσουμε βάρος στο μέλλον και χαίρομαι για το ότι αναπέμφθηκαν αυτά τα πράγματα στην Επιτροπή θα πρέπει να δώσουμε βάση ε, στο ότι όταν μιλάμε για παραγωγούς δεν είναι μόνο τεράστιε εταιρείε, αλλά και οικογενειακές επιχειρήσεις τις οποίες ε, δεν πρέπει να τις ε, παραφορτώσουμε με νομικές φιωριτούρες. Ευχαριστώ. Όταν οι ψηφοφόροι με ρωτάνε ποιο είναι το όφελος της συμμετοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εγώ τους απαντάω το ελεύθερο εμπόριο που υπάρχει μεταξύ των χωρών και η εσωτερική αγορά προσπαθούμε να ολοκληρώσουμε. Χαίρομαι για την οδηγία αυτή για τα δικαιώματα των καταναλωτών. Την καλωσορίζω γιατί κάνει ένα έστω και μικρό βήμα προς ε, την προσπάθεια ολοκλήρωσης και συμπλήρωσης της εσωτερικής αγοράς. Θα βοηθήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και το διασυνοριακό εμπόριο ή το ηλεκτρονικό εμπόριο. Βέβαια ήταν πολύ χρονοβόρα διαδικασία ε, παρασκευής αυτής της ε, οδηγίας και η πρόοδος είναι σχετικά μέτρια. Χρειαζόμαστε ένα καλό νομικό πλαίσιο για να ολοκληρώσουμε την εσωτερική αγορά και όχι τις κατακαιρματισμένες πρωτοβουλίες ε, που έχουμε αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ. Εναρμονισμένα δικαιώματα των καταναλωτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω κατοχυρώνονται από την οδηγία αυτή, είναι πολύ σημαντικά μέτρα για την ολοκλήρωση και την εύρυθμη λειτουργία τη εσωτερική αγορά. Αυτή η εναρμονισμένη οδηγία που καλύπτει πολλές προηγούμενες οδηγίες για τα δικαιώματα καταναλωτών, θα πλουστεύσει κατά πολύ το νομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην εσωτερική αγορά. Ταυτόχρονα διευκολύνει το διασυνοριακό εμπόριο και μειώνει τον κατακαιρματισμό στην εσωτερική αγορά. Δυστυχώ, η πλήρη εναρμόνιση της προστασία των καταναλωτών δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά τουλάχιστον πραγματοποιήσαμε ένα σημαντικό ποιοτικό άλμα προς μια ενισχυμένη προστασία των καταναλωτών, και αυτό και υπέρ τη έκθεσης. Η έκθεση για στην Ιαπωνία, ο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε οι ειδήσει ε, του σεισμού από τις 11 Μαρτίου ενδιαφέρει την Απανατολή και ιδιαίτερα την Ιαπωνία όλοι μας έφασαν έκπληκτους μπροστά στο έβρος της καταστροφής, της ανθρώπινης καταστροφής. Γι' αυτό θεωρώ ότι το ψήφισμα είναι ένα πρώτο υποχρεωτικό βήμα έτσι ώστε η άμαχος πληθυσμός της Ιαπωνίας να έχει όλη την ανθρωπιστική, τεχνική και οικονομική βοήθεια που θα χρειαστούν τα επόμενα χρόνια. Αυτό που έγινε στον πυρηνικό σταθμό της Φουκουσίμα μας υποχρεώνει όλους να σκεφτούμε πάρα πολύ προσεκτικά και νυφάλια τους κινδύνους της πυρηνικής ενέργειας. Η Ευρώπη πρέπει να επενδύσει και να καλέσει τα κράτη-μέλη να ποντάρουν περισσότερο σε εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Η σχέση μας στρέφεται προς την Ιαπωνία σήμερα και η δέσμευσή μας για το μέλλον θα είναι να αποφευθούν να επαναληφθούν παρόμοια στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο. Ευχαριστώ. Uh, Πριν να δώσω το λόγο στον κύριο Ρούμπικ, θα ήθελα να υπενθυμίσω στους ευρωβουλευτές ότι όταν θέλουν να υποβάλουν επεξηγήσεις πηλήφθη θα πρέπει να το... θα ενημερώνουν την γραμματεία εκ των προτέρων. Δεν είναι διαδικασία ΚΑΤΣΔΙ. the δίνω το λόγο κύριε Ρούμπικ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω πως η κατάσταση αυτή μας οδηγεί σε κάποια διδάγματα και ειδικά όσον αφορά τα πυρηνικά εργοστάσια και ζητώ από το Συμβούλιο να καταθέσει επιγόντως προτάσεις. Αυτά τα οποία έχει υποβάλει μέχρι στιγμής η Κομισιόν είναι ερέθισμα έτσι ώστε η ομάδα εργασίας πυρηνικής ενέργειας του Συμβουλίου να ανταποκριθεί επιτέλους στις απαιτήσεις του Κοινοβουλίου. Χρειάζεται μια εντατική συζήτηση και έχει φτάσει η ώρα να γίνει αυτή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, έχω λάβει από τον ε, κύριο Λουίτζι Ντε Μάτζιστρη αίτηση προάσπιση τη ασυλία του και των προνομίων του στο πλαίσιο δικαστική δίωξη που εκκρεμεί ενώπιον του δικαστηρίου του Καταντζάρο. Σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφο 3 του κανονισμού, η έτσι παραπέμπεται στην αρμόδια Επιτροπή Νομικών Θεμάτων.